κύρωση ε, ε, δόθη και ισχύουν οι εντολές αυτές. Από την αρμόδια ομάδα έχω ε, αιτήματα από αρμόδιες ομάδες για τους διορισμούς σε επιτροπές και αντιπροσωπείες. Αν μέχρι την έγκριση των πρακτικών δεν θα υπάρξει κάποια ένσταση, θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται αυτοί οι διορισμοί. Η διάσκεψη των Προέδρων, κυρίε και κύριοι, έχει τις εξής προτάσεις για την διεξαγωγή